παρά του αποκεντρωμένου δυστικού οργανισμού, το ποσό θα ευθυγραμμιστεί με την απόφαση τη Κομισιόν του Ιουλίου 2013. Για τη γάμο περιβάλλον κλίμα, συμφωνούμε με την έκθεση και με τα σχόλια των βουλευτών. Υπάρχει εστίαση στην ε, απόδοση, στις επιδόσεις, αλλά ίσως η εστίαση στην απασχόληση και στην ανάπτυξη θα μπορούσε να πάει σε διαφορετική κατεύθυνση από ότι σε σχέση με του περιβάλλοντικούς στόχους, αλλά θα συνεργαστούμε με του συναδέλφου μα για να το αποφύγουμε αυτό. For Κατά τα λοιπά, και εμεί θεωρούμε ότι το 2016 η κατάσταση για τι επιστώσεις πληρωμών θα είναι καλύτερη. Κυρίως γιατί αναβλήθηκε και δρομολόγηση κάποιων προγραμμάτων και το 2016 θα ξεκινήσει ενδιάμεση αξιολόγηση. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε αποτελέσματα και να δρομολογηθούν διάφορα project για να μπορέσουμε να τα αξιολογήσουμε σε αυτή τη διαδικασία. Σαν πρόεδρο, ευχαριστώ πολύ. Με χαρά άκουσα ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα σε τέτοιε πληρωμές. Αν όμως αργότερα ακούσω ότι δεν έχουμε πρόβλημα γιατί απλά αναβάλαμε κάποια προγράμματα. Ε, τώρα μετά αλλάζει η άποψη που, και η χαρά μου. Ε, μετριάζεται. Γιατί εμείς αυτό που θέλουμε είναι να αυξηθούν οι πόροι μας ό,τι αφορά τις πληρωμές. Γιατί μπορεί κανείς να κλείσει το προπλήσμα με δύο τρόπους, είτε με την αναβολή ε, πληρωμών, είτε με αύξηση του προβλεπόμενου πόσου. Εμείς θέλουμε να αυξήσουμε, όχι να αναβάλουμε. Εσείς λέτε τώρα ότι τελικά με αναβολή πληρωμών γίνεται αυτό, αλλά αυτό δεν είναι η προτεραιότητά μας στο Κοινοβούλιο, όπως γνωρίζετε τέλος πάντων. Σας ευχαριστώ και τώρα να σας θυμίσω το χρονοδιάγραμμα. 26 Μαΐου λίγη προθεσμία κατάθεση τροπολογιών. Στην Επιτροπή ΕΝΒΙ ψηφίζουμε 16-17 Ιουνίου και στην Επιτροπή Προπολογισμών 22-23 Ιουνίου. Και τώρα μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο. Συνέχεια της πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών Right to Water. Έχει συνταχθεί σχέδιο έκθεσης από τη συνάδελφο Λίν Μπόιλαν, στην οποία και θα δώσω αμέσως το λόγο. Κυρία Μπόιλαν, λοιπόν, έχει το λόγο για να μας εξηγήσει το ε. περιεχόμενο της έκθεσής της. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη γιατί αυτό που θέλω ουσιαστικά να ακούσω τις ε, απόψεις των σκιωδών και των λοιπόν συναντέλφων για το σχέδιο έκθεσης θα ξέρετε ότι φυσικά το δικαίωμα είναι στο νερό ε, είναι ένα δικαίωμα και η το Μάιο του 2012 ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία, πέρασε το 1 εκατομμύριο υπογραφών και σχεδόν διπλασιάστηκε 1,9 εκατομμύριο υπογραφές συνελέγησαν συνολικά. Ήταν η πρώτη μεγάλη τέτοια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία. Η παροχή νερού, η διαχείριση νερού φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα για τους πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο μηχανισμός αυτός είχε χαιρετηθεί από την Επιτροπή ως ένα μέσο για την συμμετοχική δημοκρατία που θα παρήχε μια πλατφόρμα για τους πολίτες για να επηρεάζουν, να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων, στη διαδικασία αυτή. Αλλά ε, δυστυχώς τελικά δεν φαίνεται να τηρούνται όλες αυτές οι υποσχέσεις. Αυτή η ε, πρωτοβουλία ε, θα είχε ως αποτέλεσμα να πρέπει να προτείνει η Κομισιόν νομοθεσία για να καθιερώνει το δικαίωμα στην ε, γηνή, στην υδροδότηση για υγειονομικές, μάλλον για υπηρεσίες ύτρευσης αποχέτευσης, καθολική πρόσβαση στο νερό και την υγιεινή το θετικό είναι ότι με βάση αυτή την εκστρατεία η Κομισιόν αφαιρεί από την οδηγία περί συμβάσεων παραχώρησης στο νερό και την υγιεινή, όπως επίσης ε, και το ότι υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση ό,τι αφορά την απελευθέρωση των ε, υπηρεσιών υδροδότησης. Υπήρξε μεγαλύτερη προβολή, λοιπόν, δημιουργήθηκε μια πλατφόρμα διαλόγου για το πώς επηρεάζει, μπορεί να επηρεάσει απελευθέρωση ε, τους πολίτες. Και όπως είπαμε και θέλουμε να ενισχυθεί και το δικαίωμα για την παροχή νερού σε όλη την Ευρώπη. Όμως το αποτέλεσμα οι διοργανωτές το θεώρησαν απογοητευτικό και υπογράφοντας βέβαια την πρωτοβουλία γιατί δεν δεσμεύτηκε η Κομισιόν να προχωρήσει σε νομοθεσία που θα αναγνωρίσει το δικαίωμα στο νερό σαν ανθρώπινο δικαίωμα. Είναι ανησυχητικό αυτό. και για την ίδια τη φήμη της πρωτοβουλίας αυτής, γιατί αν οι ηγέτες ένωση θέλουν πραγματικά να αποδείξουν ότι είναι δεσμευμένοι ε, στον εκδημοκρατισμό του πολιτικού θεματολογίου και αν θέλουν να ακούνε τη φωνή των πολιτών, δεν πρέπει να δίνουν τέτοιες αδύναμες απαντήσεις και αποκρίσεις. Ε, αυτός ο ενιαίος μηχανισμός δεν πρέπει ε, να γίνει όλο και πιο ασήμαντος. Γι' αυτό θα πρέπει να έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Γι' αυτό στην έκθεσή μου ζητώ πιο συγκεκριμένη δέσμευση για νομοθεσία μετά από κατάθεση μιας τέτοιας πρωτοβουλίας. Ευρωπαίων πολιτών. Μέχρι στιγμής ε, η Κομισιόν ήταν υπέρ μιας προσέγγισης ε, που βασίζεται στον ε, ανταγωνισμό της υπηρεσίας αγοράς, απελευθέρωση υπηρεσιών στον τομέα της ίδρυυσης και δεν αναγνωρίσει τόσο το ρόλο των δημόσιων κοινοφιλών υπηρεσιών. Εγώ εφιστώ την προσοχή στο ότι η παροχή του νερού είναι ένα εθνικό μονοπόλιο δεν μπορεί να είναι αποτέλεσμα ανταγωνισμού στις αγορές και όπου έχει υπάρξει η απελευθέρωση της ιδιοκτησίας βλέπουμε πολύ λίγα να επανεπενδύονται στις ε, υποδομές ε, ίδρευσης. Υπήρξε μια τεράστια, μια φανταστική υποστήριξη αυτής της πρωτοβουλίας. Και βλέπουμε ότι οι πολίτες δεν συμφωνούν ότι έχει νόημα απελευθέρωση των υπηρεσιών ε, ίδρυυσης. Από πολλές χώρες ε, οι πολίτες από την Ιρλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ισπανία κτλ. Λένε όχι σε αυτές τις ε, διαδικασίες απελευθέρωσης, ε, τονίζω την πρωτοβουλία των Παρισίων. Και επίσης κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει είναι η συντήρηση, η διατήρηση των πόρων. Έχουμε όλο και πιο μεγάλη σπάνιδα πόρων. Η σημασία του νερού ως φυσικού πόρου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Επίσης εκπαίδευση για τη διατήρηση του νερού. Νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση αυτό και στην οδηγία πλαίσια για τα ύδατα και όχι μόνο για την ε, χώρα κατανάλωση, την κατανάλωση στην οικιακή μάλλον, αλλά και στον γεωργικό τομέα, γιατί ο τομέας αυτός χρησιμοποιεί τεράστιες ποσότητες νερού. Επίσης θα ήθελα να περιληφθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ανάγκη μετώπισης της ρήπανσης ε, στην πηγή. Είναι καλύτερη πρόληψη παρά να εξεργαζόμαστε, να ε, καθαρίζουμε το νερό μετά. Θα υποβάλω περαιτέρω τροπολογική και στη δική μου έκθεση για να επεκταθώ περισσότερο σε κάποια από τα θέματα που σας προανέφερα και ελπίζω ότι θα συνεργαστούμε αποδοτικά και επικοδομητικά και με τους συναδέλφους. Με ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα γίνει ο πρώτος γύρος. Η κυρία Ράνς η πρώτη. το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την συνάδελφο. Έχουμε διαβάσει την εκθεσή σας και θα ήθελα να σας πω ότι εν γέννη Αναγνωρίζω ότι η πρωτοβουλία Ευρωπαϊκών Πολιτών είναι μια καλή πρωτοβουλία. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι οι πολίτε πρέπει να μπορούν να απευθύνονται άμεσα στο Κοινοβούλιο και να προωθούν την δημιουργία νομοθεσία. Από εκεί και πέρα βέβαια το να δώσουμε σε αυτή την πρωτοβουλία την εξουσία να μπορεί να τροποποιεί ε, θέσεις της Κομισιόν για κάποια κείμενα τα οποία τα περιλαμβάνετε σε μια παράγραφο της έκθεσής ε, σας είναι λίγο μακριά, ε, έχει μια μεγάλη απόσταση και να μην, είμαστε, να μην θριαμβολογούμε ε, τόσο νωρίς. Υπάρχουν δύο-τρία σημεία τώρα για να συμπληρωθεί η εκθεσή σας. Το πρώτο, η σχέση της νομοθεσίας και πόσο ε, η διεθνής νομοθεσία μπορεί να επηρεάσει Υπάρχουν κάποια ψηφίσματα, πούμε, το τελευταίο των μέθων. δεν το συμπεριλαμβάνεται. Μια ανάπτυξη του 2013 συγκεκριμένα, πολύ σημαντικό. Επίση, κάποια σύγχυση μεταξύ ε, τη Γενική Συνέλευση των Εθνών και τη Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τα μπερδεύεται αυτά τα δύο. Το Συμβούλιο, μάλλον, των Δικαιωμάτων έχει λάβει πολύ σημαντικέ αποφάσει. Θέλω να καταθέσω με τροπολογία. Πρώτον, περιλαμβάνω το, πρώτο το τελευταίο ψήφισμα των ΟΕΦ και δεύτερον, Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Γιατί το δικαίωμα στο νερό το αναγνωρίζει η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Δεν έχει ψηφιστεί από τη Γενική Συνέλευση των ΕΕ ακόμη. Να μην λέμε λοιπόν ότι έχει αναγνωριστεί από τη Γενική Συνέλευση είναι ψέμα. Να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι όταν λέμε τι έχει εγκριθεί και τι δεν έχει εγκριθεί ακόμα από τα Ηνωμένα Έθνη. Σε ένα διαφορετικό επίπεδο. Πολύ σημαντικές οι αναφορές στον εισηγητή και στην εισηγήτρια κατά το παρελθόν, το να για το νερό. Η προηγούμενη εισηγήτρια Κατερίνα Δεαλμπουκέρκη είχε κάνει κάποιες εκθέσεις ε, και κάποιες παρατηρήσεις ε, που ε, παραμένουν επίκαιρες. Η κυρία Κατερίνα Αλμπουκέρκη, η προηγούμενη λοιπόν εισηγήτρια, είχε γράψει πολύ ξεκάθαρα ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός δημόσιου αγαθού που Άλλο τώρα αυτό, αν θα το διαχειρίζεται αυτό το δημόσιο αγαθό, μια δημόσια ιδιωτική επιχείρηση. Και έλεγε ότι οι συμβάσει παρακόρηση των Δήμων είναι θεμητέ. Επομένω, νομίζω ότι αναφορά στον εισηγητή σε αυτό το έγγραφο είναι πολύ σημαντικό ε, στοιχείο και γι' αυτό θα καταθέσω εγώ τροπολογίε. Επίση, μα βλέπετε εκφράζεται κάποιε ανησυχίε για τη διαχείριση. Μα ε, την ευθύνη την έχουν οι Δήμοι οι Δήμοι, η τοπική αυτοδιοίκηση έχουν. Ε, πρέπει να λάβουν τι αποφάσει για τη διαχείριση. Μπορεί να δημιουργηθεί μια δημόσια επιχείρηση που θα πάρει αυτή τη σύμβαση παραχώρηση. Ή μπορεί να αποφασίσει ένα Δήμο να ε, έχει ένα συμβόλαιο με μια ιδιωτική επιχείρηση. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ συγκεκριμένοι, πολύ λεπτομερείς. Έχουμε το 345 άρθρο που λέει πρέπει να είμαστε αμερόληπτοι, αντικειμενικοί. Άρα πρέπει να σεβόμαστε την νομοθεσία, τη δική μας νομοθεσία της Ένωσης. Και για τα 28 κράτη μέλη. Επίσης να σας πω ένα παράδειγμα από τη χώρα μου. 50% ή 60-40 ή δεν ξέρω αν είναι 43-57. Έχουμε διαρρέσει έτσι τέλος πάντων ε, τους Δήμους που έχουν διαχείριση από δημόσιες ή από ιδιωτικές. Υπάρχουν ε, παραδείγματα πολύ καλής διαχείρισης και δεν έχει καμία σχέση αυτό με τα πολιτικά χρώματα ή κόμματα. Έχουμε κάποια διαχείριση από αριστερούς δήμους με ιδιωτικές επιχειρήσεις και έχουμε κάποιους δεξιούς δήμους ή κεντρώους που έχουν ε, δημόσιες ιδιωτικές Δεν είναι καθόλου πολιτικό το θέμα, είναι θέμα κοινή λογικής. Πώς θα παράσχουμε μια ε, αξιοπρεπή αποτελεσματική υπηρεσία στους πολίτες με το μικρότερο δυνατό κόστος. Και θα περάσω τώρα σε μια άλλη για το κόστος, στην τιμή. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα είδος ε, εξεταστεί, αν θέλετε, ε, που μια, μια τέτοια μορφή να δημιουργήσουμε, που θα ερευνά τι γίνεται. Το νερό είναι δωρεάν. Αυτό που δεν μπορεί να είναι ε, δωρεάν όμως είναι ε, η υδροδότηση, οι σωληνώσεις, ο καθαρισμός, ο βιολογικός στη συνέχεια, και η συνεχή βελτίωση τη παροχή αυτή τη υπηρεσία. Άρα νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δημιουργήσουμε αυτόν τον λεγόμενο εξεταστή, ένα άτομο ή τέλο πάντων ένα φορέα εθνικό, εγώ θα καταθέσω σχετικά τροπολογίε που θα είναι αρμόδιο και ο οποίο θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να ερευνά, να επιθεωρεί ότι παρέχουν όλοι οι Δήμοι την απαιτούμενη υπηρεσία και θα διευκρινίζει τι πληρώνει, τι πληρώνει με την, το τιμολόγιο του νερού πολίτης, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Τι πληρώνουν ακριβώς όταν πληρώνουν το λογαριασμό του νερού. Και θα υποβάλω και μία τροπολογία πάντα σε αυτό το πλαίσιο. Γιατί αναγνωρίζω ότι έχετε δίκιο σε έναν βαθμό. Μιλάτε για την οικονομική κρίση. Αλλά και πριν από την οικονομική κρίση, πάντα υπήρχαν ομάδε του πληθυσμού που βρίσκονταν σε δύσκολη, σε ευάλωτη θέση και αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να έχουν πρόβλημα. Να πληρώσουν το ρεύμα, το νερό, ε, το φυσικό αέριο, οτιδήποτε άλλο. Πρέπει όμως να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν ε, μέρη όπου λειτουργεί ήδη ένα αποτελεσματικό σύστημα κοινωνικής προστασίας και ασφάλεια. Πάλι εδώ δίνω παράδειγμα από τη χώρα μου την Ισπανία που έχουμε μια τέτοια ε, μορφή. Αν δηλαδή σε ένα δήμο ένα νοικοκύριο δεν μπορεί να πληρώσει το νερό, τι γίνεται, ο δήμος αναλαμβάνει να πληρώσει το λογαριασμό ή η ιδιωτική ιδιωτικη εταιρεία. Διαβιβάζει στο Δήμο το πρόβλημα και οι κοινωνικές υπηρεσίες που εγγυώνται ακριβώς ότι περί αυτού πρόκειται και όχι, δηλαδή περί αδυναμή και όχι περί απάτης. Γιατί αν μιλήσετε λίγο με τους παρόχους υπηρεσιών και ιδιωτικούς και δημόσιους παροχής ε, υπηρεσιών γραβδότησης, υπάρχει, θα σας πω ότι υπάρχουν πολλοί που σταματά να πληρώνουν γιατί αλλάζουν σπίτι αλλά δεν ενημερώνουν ότι μετακόμισαν ή ε, κλείνει μια επιχείρηση, αλλάζει την έδρα της κτλ. Ή γιατί δεν θέλουν να πληρώσουν πολύ απλά, υπάρχουν και αυτοί. Για να μην έχουμε λοιπόν ε, ανοίξει μια πόρτα που να μπορεί να περνά ποιος θέλει από εκεί, υπάρχει αυτή η μορφή, αυτή η αρχή. Και αυτό μπορεί να αποτελέσει, πιστεύω, παράδειγμα παρασμένες και από άλλες χώρες. Γιατί είναι καλό να υπάρχει αυτή η κοινωνική υπηρεσία για το νερό. Τέλος, να σας πω ότι εγώ νομίζω ότι γέννη είναι ενδιαφέρον να έχουμε υπόψη την ανησυχία που μπορεί να προκύψει, όπως στη χώρα μου, στην ακτή του Λεβάντε. Ε, μπορεί να προκύψει πρόβλημα και ανησυχία με τον νερό. Υπάρχουν κράτη-μέλη, πρέπει να τον αναγνωρίσουμε και λυπάμαι που το λέω. Που επειδή είχαν πολύ νερό πάντα, δεν τους ενδιαφέρει το νερό και δεν έχουν επενδύσει στο νερό. Όμως τα ωφέλη τα κέρδη που έχουν με τις ποσοστώσεις που πληρώνουν οι χρήστες, αυτά πρέπει να επανεπενδύονται συνεχώς στη βελτίωση του δικτύου. Και θα πρέπει να τραβήξουμε το αυτή στα κράτη-μέλη εκείνα που δεν έκαναν τίποτα για να βελτιώσουν το σύστημα ε, παροχής, ε, της ολυνώσης, ε, το βιλικό καθαρισμό που έχουν μολύνει τον υδροφόρο ορίζοντα. Και ερχόμαι να σας πω και κάτι ακόμη. Στη δική μου τη χώρα, την Ισπανία, πράγματι υπάρχει ανησυχία. Γιατί έχουμε πρόβλημα, έχουμε λειψιδρία. Αλλά με μια υπηρεσία που την διαχειριζόμαστε με μια συγκεκριμένη ιεραρχία και με μια συγκεκριμένη δομή, κάπως το σώζουμε, σώζουμε την κατάσταση. Όμως το θέμα δεν αφορά ένα συγκεκριμένο οικονομικό τομέα, αλλά είναι για θέμα γενικής παιδείας. Ε, πριν από κάποια χρόνια ε, πλέναμε τα δόντια μας χωρίς να κλείνουμε τη βρύση καθόλου, να αφήναμε να τρέχει συνέχεια. Τώρα, ε, για βάλτε ένα παιδί ε, κάτω των 15 να κλείνει τα δόντια του. Όλοι κλείνουμε το νερό όταν πλένουμε τα δόντια μας. Δεν το έχουμε συνέχεια να τρέχει. Έχει αλλάξει η νότροπη, έχει αλλάξει η κουλτούρα. Αυτά λοιπόν θα καταθέσω τι τροπολογίε. Το συγγνώμη που μακρηγόρησα τόσο πολύ. Είναι μια έκθεση όμω που τη μελέτησα πάρα πολύ προσεκτικά. Ε, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Και ένα τελευταίο. Αυτοί που υπέγραψαν την πρωτόβουλα δεν ήταν 1,9 εκατομμύρια, 1,6 εκατομμύρια. Αυτό λέει σε επίσημε ιστοσελίδε τη Κομισιόν. Ευχαριστώ. Και γι' αυτό θα καταθέσω τροπολογία. Ευχαριστώ, Έστερ. Είναι συγκαρσία. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, θέλω πρώτα απ' όλα να συγχαρώ την εισηγήτρια για την έκθεση της. Είναι ένα κείμενο που πιστεύω πραγματικά ακροάζεται, αφουγκράζεται αυτά που έχει προτείνει η ε, Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών και ε, αυτό δεν το έκανε δυστυχώς η Κομισιόν στο κείμενό της. Ε, Στην ανακοίνωση επαναλαμβάνονται κάποιες δεσμεύσεις. Αν με επιτρέπει κυρία Μπόιλαν να πω ότι πραγματικά είναι λίγο αποκαρδιωτικό το ότι η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών έχει αυτή την τόσο ασαφή και λίγο φιλόδοξη ανταπόκριση. Πραγματικά συμφωνώ με την ισχύ, θα πρέπει να υποτεθεί μια νέα πρόταση που δεν θα αναμασά οδηγίε όπω αυτή για τα πόσιμα ή για τα ιταλήματα. Έχουμε την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα που είναι πυλώνα τη νομοθεσία μα. Δεν μπορεί να περιοριστεί να λέει ότι δεν είναι εμπορικό αγαθό όπω τα υπόλοιπα το νερό, γιατί ε, είναι δικαίωμα το νερό. Αυτή εξ εμπόρευμα δεν ε, έχει στόχο τη δημιουργία ε, κέρδους, πλούτου σε μία από τις πιο εμβληματικές της ε, ε, οδηγίες δεσμευτικά ε, και με τα ίδια λόγια που έχουν χρησιμοποιήσει οι πολίτες στην πρωτοβουλία τους. Θα πρέπει να λέει ότι θα ε, τα κράτη-μέλη για να μπορούν να ασκούν όλοι οι πολίτες το δικαίωμά τους στην υδρότηση και στην αποχέτευση. Επίσης, μέτρα κατά της στόχιας που σχετίζεται με το νερό, την πρόσβαση του νερού, την ποιότητα του νερού. Στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει πολλά στοιχεία για, ε, ε, για το νερό, για τις αναπτυγμένες χώρες όμως, αλλά φαίνεται να παραγνωρίζει ότι εδώ στην Ευρώπη δημιουργήθηκαν μεγάλα προβλήματα ε, σε οικογένειες και σε νοικοκυριά έχουν πρόβλημα. Κόπηκε το νερό σε πάρα πολλές οικογένειες. Το ξέρει αυτή η Κομισιόν. Ξέρει ότι έχουμε πραγματικά εξώσεις ή έχουμε ε, τρομερά προβλήματα με την υδροδότηση. Θα θέλαμε να ρωτήσουμε τώρα την εισηγήτρια σε σχέση με μια πτυχή που μπορεί να δημιουργεί κάποια σύγχυση στην αρχική έκθεση. Σε κάποιες αναφορές, διατυπώσεις, ε, μπερδεύει κάπως την κυριότητα με τη διαχείριση του δημοσιογραφού. Εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να είναι σε αυτό δημόσιο ε, το νέο θέλουμε να προωθήσουμε δημόσια διαχείριση, μορφές συμμετοχικές, διαφανής και μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ε, θα μπορούσε να υπάρχει δυνατότητα παραχώρησης κάποιων στοιχείων ε, της παροχής του νερού σε, στον ιδιωτικό τομέα, πάντα με τρόπο που θα είναι απόλυτα ρυθμισμένος, καθαρισμός, το είπε και η κυρία Ράντ, στην τοπική αυτοδείξη που κάποιες φορές έχουμε δημόσια διαχείριση ή υπάρχει μια συμβάση παραχώρηση, μια ιδιωτική πτέρια, όπως και αν έχει όμως, πρέπει να εγγυηθούμε το δημόσιο χαρακτήρα του νερού και ότι ελέγχεται η διαχείριση. Πρέπει επίσης να διακρινίσουμε ότι και ο έλεγχος του πορού αυτού είναι αμετάκλητα δημόσια, αλλά θα πρέπει να γίνεται η βέλτιστη δυνατή διαχείριση ανάλογα με το μέρος, ανάλογα με το χώρο. Δεν, δεν μιλάμε για ένα εμπόρευμα που δεν είναι, δεν είναι ε, κερδοσκοπικό ε, στο χαρακτήρα της παροχής νερού. Εγώ θεωρώ ότι δημόσια πρέπει να είναι διοίκηση, όταν το βλέπουμε και στους πιο πολλούς δήμους, πώς θα και να προσανατολίζονται. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία, θα προσπαθήσω να καταθέσω τροπολογίες για κάποιες άλλες παρατηρήσεις. Εμείς θα πρέπει στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να εργαζόμαστε στα μάτια για να είμαστε κοντά ε, στην, ε, στον Ευρωπαίο πολίτη που ε, παίρνει απόσταση, αποστασιοποιείται και θα αποστασιοποιηθεί ακόμη περισσότερο αν στρίψουμε την πλάτη μας σε αυτή την πρώτη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία. Γι' αυτό είμαστε εδώ όμως, όχι για να διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια αποστασιοποίηση και μια απογοήτευση, αλλά για να εργαστούμε όπως μας το ζητά και αυτή η πρωτοβουλία. Σε ό,τι αφορά τις τιμέ θα καταδεχθούν τροπολογίες. Εγώ πιστεύω ότι με βάση το τι προβλέπει η οδηγία πλαίσιο θα πρέπει να έχουμε συστήματα όπου η ανάκτηση του κόστους θα είναι ο κεντρικός άξονας και κυρίως πρέπει να έχουμε δίκαια, ε, διαφανή, επαρκή συστήματα τιμολόγηση για να εμπιόμαστε ε, και την ποιότητα της υπηρεσίας αλλά και την παροχή της όλους τους πολίτες. Έχουμε αυτά τα θέματα για την κυριότητα και το δημόσιο χαρακτήρα του νερού, αλλά θα πρέπει και άλλα θέματα να περιλαμβάνονται στην έκθεση εξυγχρονισμός, βελτιστοποίηση υποδομών, η αποταμίευση, η εγκάρσια ζητήματα να είναι τα ζητήματα του νερού, άρα ενταγμένα σε όλες τις πολιτικές, δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας, βιώσιμη χρήση του νερού ως ανανεώσιμης πηγής ενέργειας. Πολύ δουλειά έχουμε μπροστά μας αν θέλουμε να δώσουμε στην Κομισιόν ένα σαφές μήνυμα. Και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αν θέλουμε να στηρίξουμε αυτή τη νέα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία με την οποία πιστεύω ότι όλοι συμφωνούμε το νερό. Είναι θέμα δικαιοσύνη, είναι δικαίωμα. Η πρόσφατη οικονομική κρίση το έθεσε σε κίνδυνο. Γι' αυτό πρέπει να στήσουμε να αναγνωριστεί ω δικαίωμα στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Αυτό έχει όλο και μεγαλύτερη σημασία. Σήμερα περισσότερο από ποτέ. Thank you very much, Mr. Dorman. Στο Ντόρμαν Ευχαριστώ. Συμφωνώ με το θέμα αυτό για την υγεία και για το νερό. Το αναγνωρίζουν τα κράτη-μέλη και θεωρούν ότι είναι προϋπόθεση απαραίτητη για τη ζωή και η σωστή διαχείριση των υδατίνων πόρων ε, εξασφαλίζεται μέσω της σωστής χρήσης των υδάτων στην Ευρώπη. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι καλή αυτή η επαφή, να υπάρχει επαφή με τους πολίτες μέσω της πρωτοβουλίας πολιτών. Γνωρίζουμε ότι οι πολίτες στις διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένης Πορτογαλίας, Ισπανίας, Ιρλανδίας και Γερμανίας, ανησυχούν για την φιλελευθεροποίηση στον τομέα των υδατίνων πόρων. Στην ομάδα μου θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πρέπει να προτείνει νομοθεσία σχετικά με το δικαίωμα στο νερό. Δεν νομίζουμε ότι αφορά την αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνώ με την εισηγήτρια ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να λέει ότι η ιδιωτικοποίηση θα επιβάλλει αποφάσεις στα κράτη-μέλη. Θα πρέπει η τοπική αυτοδίκηση να αποφασίζει, αυτή που είναι πιο κοντά στους πολίτες. Η πολιτική για το νερό θα πρέπει να παραμείνει στα χέρια των κρατών μελών δεν χρειάζεται να υπάρχει πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την δυτικοποίηση των τετίνων πόρων. Η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να επιβάλλει απαιτήσει σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που πρέπει να ανταποκρίνουν τις απαιτήσει τοπικής αυτοδιοίκησης. Στη Δανία υπάρχει μία αρχή ότι δεν μπορείς να βγάζεις κέρδος παρέχοντας νερό. Πρέπει να είναι, προτεραιότητα έχει ασφαλής εφοδιασμό σε νερό. Κάποιοι πιστεύουν ότι πάροχοι ύδατος βγάζουν εύκολα κέρδη και οι πολίτες την πληρώνουν τελικά. Πώς εξασφαλίζουμε ότι τα υπόγεια ύδατα που είναι σπάνια δεν καταστρέφονται με τη λάθος μεταχείριση και ότι δεν υπάρχει υπεράσπιση ε, συμφερόντων απλευράς εκείνων που χειρίζονται τους ε, υδάτινους πόρους ε, προσβλέπω σε συνεργασία ε, και θα θέλουμε να εξασφαλίσουμε στους πολίτες ότι θα έχουν καθαρό νερό στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φαρία έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ την συνάδελφό μου τη Λίν Μπόιλαν. Έκανε πολύ καλή δουλειά όσον αφορά το σχέδιο εκθέσεως. Η ευρωπαϊκή αυτή πρωτοβουλία πολιτών για το δικαίωμα στο νερό έχει τρεις στόχους. Πρώτον, Ευρωπαϊκή Ένωση κράτη-μέλη να έχουν υποχρεώσει να εξασφαλίζουν ότι όλοι οι κάτοικοι απολαμβάνουν το δικαίωμα στο νερό και ε, στην ε, υγεία. Και δεν θα πρέπει να αποκλείονται όμω η υδάτινη πόρια από την απελευθέρωση και θα πρέπει να υπάρχει καθολική πρόσβαση στο νερό και στην ε, αποχέτευση. Χρειάζεται σωστή διαχείριση των ε, δατίνων πόρων και το μοντέλο της ιδιοκτησίας αφορά την επικουρικότητα και μπορούν να επιλέξουν το θέμα αυτό τα κράτη-μέλη. Η έκθεση τι αναγνωρίζει. Διαφοροποίηση του νερού από άλλα αγαθά. Να θεωρείται δημόσιο αγαθό και ανθρώπινο δικαίωμα για να υπάρχει καθολική πρόσβαση σε επαρκείς ποσότητες καθαρού νερού για προσωπική και οικιακή χρήση πρέπει να έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία, να γίνουν σωστές επενδύσεις, σωστοί μηχανισμοί διαχείρισης, βιώσιμη διαχείριση του νερού και από πλευράς οικονομικής και περιβαλλοντικής. Ανεξάρτητα το μοντέλο που θα επιλεχθεί από το κάτω μέλος, πρέπει να εξασφαλίζουμε ότι θα οδηγεί σε χαμηλές τιμές, κυρίως για τους φτωχούς. Να είναι αποδοτική η χρήση των υδατίνων πόρων και τα διάφορα οικοσυστήματα προστατεύονται. Χρειάζεται περισσότερες επενδύσεις για τεχνολογική εξέλιξη και καινοτομία. Εκπαίδευση, παιδεία. Να αλλάξει ο τρόπος χρήσεως των υδατίνων πόρων. Μεγαλύτερη διαφάνεια, συμμετοχή των καταναλωτών, μεγαλύτερος έλεγχος των διαφόρων επιχειρηματικών μοντέλων ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών, βαθμολόγηση αυτών και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Και θα πρέπει και οι δύο τομείς να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων. Χρειάζεται ανεξάρτητη αρχή ελέγχου διαχείριση των υπερτείνων πόρων. Πρέπει να προστατεύουν τα συμφέροντα των καταναλωτών οι φορεί αυτοί. Όπω είπε ο συνάδελφο από το ΕΛΚ, χρειαζόμαστε ανεξάρτητο φορέα, έναν κάποιον που προστατεύει τους καταναλωτές του ύδατος και να απευθύνονται σε αυτό το πρόσωπο ε, οι πολίτες για προβλήματα. Ένα είδος διαμεσολαβητή για το νερό. Χρειάζεται μεγαλύτερος ρόλο στις ρυθμιστικές αρχές για το νερό, καλύτερη συνεργασία μεταξύ τους. Έτσι βελτιώνονται οι πρακτικές και θα γίνει ανταλλαγή γνώσεων. Καινοτόμε δύσεις πρέπει να θετούνται τάχιστα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί ο μονοπωλιακός χαρακτήρας των υπηρεσιών νερού. Κάποιες πρωτοβουλίες διαμορφώνονται και πρέπει να στηριχθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα προτείνω τροπολογίες σχετικές. Προσβλέπω σε συνεργασία με τους συναδέλφους. Και με την εισηγήτρια και τους πιο εισηγητές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και κύριος Λαφρόντι από την ε, ομάδα FTD. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ την εισηγήτρια. Αξιοσημείωτη η εργασία που έκανε, λεπτομερέστατη, διευκολύνει τις εργασίες μας. Έχει διαιρεθεί έκθεση σε τμήματα, σε κομμάτια ανάλογα με τα επιχειρήματα. Με λογική προσέγγιση. Το εκτιμώ αυτό και κάποια από τις ομάδες των θεμάτων αφορά την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Όχι που συνδέεται με το right to water, αλλά σαν ένα μέσο άμεσης δημοκρατίας των πολιτών. Δυστυχώς δεν έχει λειτουργήσει όπως θα έπρεπε. Λέμε στους πολίτες ότι μπορούν να συμμετάσχετε και να απευθύνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν συλλέξετε ένα εκατομμύριο υπογραφές, όταν συλλεχθούν οι υπογραφές που απαιτείται, Στο τέλος, η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι απλώς μια ανακοίνωση. Η εμπιστοσύνη των πολιτών στους ευρωπαϊκούς θεσμούς είναι πολύ χαμηλή. Όταν κάνουν σημαντικές προσπάθειες και παίρνουν τέτοια απάντηση, η εμπιστοσύνη μειώνεται. Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι αδύναμη και στη μορφή και στην ουσία. Ζητούν τρία πράγματα οι πολίτες και η καρδιά του αιτήματος ήταν επιτέλους μια απάντηση για τη φιλελευθεροποίηση των νερών. Η απάντηση ήταν απλώς ότι αυτό είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών και θέμα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και είναι το καλύτερο μέσο, αλλά δεν αλήθεια δεν μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ασκήσει πιέσεις για να γίνουν πράγματα σε τοπικό επίπεδο. Περιμέναμε απάντηση νομοθετικού είδους. με νομοθετική πρόταση, ανταυτού έχουμε μια ανακοίνωση. Το μέγιστο που πετύχαμε. Αυτό αποτελεί απογοήτευση προφανώς έναντι των διαφόρων κινημάτων. Έγινε συνάντηση του Ευρωπαϊκού Κινήματος για το νερό στις Βρυξέλλες κάποιες εβδομάδες και έχουν σχηματιστεί πολλά κινήματα για αυτό το ζήτημα στην Ιταλία το 2011. Έγινε δημο... Κάναμε δημοψήφισμα, 27 εκατομμύρια Ιταλοί ψήφισαν για το δημόσιο νερό, 95% ναι, θέλαμε να είναι δημόσιο αγαθό το νερό, όμως η, η μεγάλη νίκη και οι γιορτές οδήγησαν σε απογοήτευση, διότι για την ώρα είμαστε πολύ πίσω όσο αφορά την υλοποίηση των αποτελεσμάτων δημοψηφίσματος. Για τα συγκεκριμένα σημεία τώρα που μπορούμε να τα επεξεργαστούμε και να υποβάλουμε τροπολογίες. Η συγγήτρια και στη συζήτηση ανέφερε, αναφέρθηκε αυτό που αναφέρει. Πολλά άτομα δεν έχουν πρόσβαση στο νερό και το φαινόμενο αυξάνεται. Δεν έχουν τα χρήματα, βλέπετε, για να πληρώσουν το λογαριασμό για το νερό. Στη χώρα μου είναι πολύ ανησυχητικό αυτό που συμβαίνει και σε άλλες χώρες. Όλο αυξάνεται αυτό ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν πρόσβαση στο νερό θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα βηματάκι παραπάνω, μια προσπάθεια θαραλέα να προτείνουμε ελάχιστη, ελάχιστη ποσότητα ύδατος εγκυμένη για κάθε πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπενθυμίζει ότι η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας δίνει στοιχεία αριθμητικά. Για κάθε πολίτη θα ήταν καλό να έχει ε, έναντι 50 με 100 λίτρα την ημέρα διαθέσιμα. Ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ποσίμου ύδατος θα μπορούσε να είναι κάτι καινοτόμο, αλλά σημαντικό, για να προστατεύσουμε ένα ανθρώπινο δικαίωμα. Κάτι άλλο. Συχνά μιλάμε για την αλλαγή του κλίματος. Δεν το θεωρούμε μόνο σαν μάχη, αλλά και ανάγκη προσαρμογής και αντοχής στην αλλαγή του κλίματος. Και χρειάζεται η προστασία του, ε, ε, του ύδατος, του πόσιμου, ε, έναντι της αλλαγής του κλίματος. πρέπει να γίνει μια προσαρμογή στις καταστροφικές συνέπειες της αλλαγής του κλίματος που σημειώνεται παντού σε όλο τον κόσμο αλλά σε κάποιες χώρες, κυρίως στις τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα καταστροφικά υπενθυμίζω κάτι που λησμονούμε είμαστε πολύ πλούσιοι στη Δύση ότι το πόσιμο νερό, το γλυκό νερό είναι άκρος περιορισμένος πόρος μόνο το 3% όλων των υδάτων του πλανήτη είναι γλυκό νερό και τα 2 τρίτα του 3% είναι φυλακισμένα στους παγετώνες. Άρα το πόσιμο νερό, μόνο 4% αυτών των υδάτων είναι πόσιμο και διαθέσιμο. Δεν είναι μόνο περιβαλλοντική μάχη, αλλά και μάχη επιβίωσης αν θέλετε, του ανθρωπίνου είδους. Σε κάποιο άλλο σημείο της εκθέσεως αναφέρεται η προστασία των φυσικών αποθεμάτων του γλυκού ύδατος και των οικοσυστημάτων του γλυκού ύδατος. Είναι θεμελιώδες να διαφυλαχθεί αυτή η σπάνια πηγή. Και πρέπει να προστατευτεί και το δικαίωμα της πρόσβασης των ανθρώπων σε αυτή την πηγή. Πρέπει να αποφύγουμε και τη σπατάλη του γλυκού νερού, του ποσίμου νερού, Χρειάζεται ευαισθητοποίηση, εκστατείες, επικοινωνία. Γίνονται πολλές προσπάθειες. Εδώ και 20 χρόνια, όπως είπε η συνάδελφος, κάναμε πολλά βήματα προόδου, αλλά από αυτή την άποψη όσον αφορά την ανακοίνωση για τη σπατάλη του ύδατος δεν αρκούν ποτέ οι προσπάθειες, γιατί και στην Ευρώπη γίνεται σημαντικότατο θέμα, πρέπει να επιμείνουμε και στην Ευρώπη πρέπει να επεξεργαστούμε τις δομές. Έχουμε σωληνώσεις για το νερό στην Ευρώπη, και το ανέφερε η Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Ευρώπης στη έκθεση, οι σωληνώσεις χάνουν τουλάχιστον 10% μέχρι 40% του νερού που μεταφέρουν. Είναι σπατάλι λόγω διαρροών. Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε αυτό και θα πρέπει οι υποδομές να βελτιωθούν για να προστατεύσουμε τόσο ευαίσθητη πηγή που είναι σημαντικότερη τον άνθρωπο. Ευχαριστώ. Η κυρία Περίκη έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, ε, θέλουμε να δώσουμε συνέχεια στην, ε, Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών για το νερό, που είναι σημαντικό σε πολλές χώρες και πάρα πολύ σημαντικό και στην Ολλανδία. Δεν είναι μόνο το θέμα του ασφαλούς ποσίμου ύδατος ε, για τους ανθρώπους, για τα σπίτια, τα νοσοκομεία, τα σχολεία. Ε, το θέμα έχει να κάνει και με την καινοτομία. Η Γεωργία τα εξετάζει αυτά. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει ευαισθητοποίηση και ενημέρωση. Μπορεί κανείς αντί να κάθεται κάτω από τον ντους 10 λεπτά μπορεί να καθαριστεί και στα 2 λεπτά. Τώρα, για το ψήφισμα για το ανθρώπινο δικαίωμα πρόσβαση σε πόσιμο νερό και αποχέτευση. Αυτό πρέπει να το υποστηρίξουμε. Αλλά αν δούμε την οδηγία πλαίσιο για το νερό, και την νομοθεσία για το πόσιμο νερό ε, είναι σωστό να ε, κατοχυρώνουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα έτσι. Όχι, αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα κατοχυρώνονται στις ε, συμβάσεις. Επίσης, το θέμα της πληρωμής των λογαριασμών ύδατος δεν έχει να κάνει με κάποια, κάποιο φταίξιμο της εταιρεία ίδρευσης, αλλά ε, φταίει η κρίση που θυματοποιεί τους πολίτες. Πρέπει λοιπόν να δούμε επίσης και τις συμπράξεις μεταξύ δημοσίου αλλά και με ιδιώτες και να δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε δυνατότητες για να επιτύχουμε το στόχο του καθαρού νερού. Ε, τώρα, το Ταμείο Αλληλεγγύης για το νερό και οι κοινωνικοί κανόνες, αυτό πρέπει να παραμείνει στα χέρια των κρατών μελών. Ε, υπάρχει επιμερισμένη ευθύνη. Νομίζω στη χώρα μου υπάρχουν αρκετοί ε, κοινωνικοί κανόνες ήδη για τους πολίτες. Ευχαριστώ τώρα η κυρία Ντελχάγη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στρέφομαι στους συναδέλφους εκ μέρους και του Μισελ Ταντά και μου βέβαια ο κύριος Ντάντα δεν μπορούσε να είναι εδώ σήμερα. Η πρόσβαση στο νερό είναι ένα σημαντικό ζήτημα, μεγάλη πρόκληση για το μέλλον. Και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με άκρο ρεαλιστικό τρόπο αυτό το ζήτημα. Θα πρέπει επίση να μα απασχολήσει και το ζήτημα τη πέτρας και το ζήτημα τη ποσότητα, και θα πρέπει να το δούμε όλο αυτό υπό το πρίσμα των επιπτώσεων που έχει αλλαγή του κλίματο. Κάτι που δεν αποτελεί πια υπόθεση σήμερα, αλλά πραγματικότητα. Ποσότητα νερού για τη διατήρηση και λέω διατήρηση ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων, όχι μόνο γεωργικών αλλά και για τη βιομηχανία. Είναι ένα πάρα πολύ οξύ πρόβλημα, όπως είναι και ε, το θέμα της πρόσβασης του πληθυσμού σε επαρκές νερό, ποιοτικό νερό. Θα πρέπει να μας απασχολήσει το ζήτημα του νερού σε κοινωνικό επίπεδο, ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών καθαρισμός του νερού πριν και μετά την οικιακή χρήση. Όλα αυτά δίνουν, ε, κάνουν το νερό πιο ακριβό και απρόσιτο σε πολλά ε, μέρη του κομματισμού που δεν έχουν τα απαραίτητου πόρους. Υπάρχουν θέματα τα οποία δεν αντιμετωπίζονται παρκώ στην ε, έκθεση. Τώρα, το θέμα δημόσιο δυτικού τομέα πρέπει να το αποδραματοποιήσουμε λίγο. Έγινε μια μελέτη πριν από κάποια χρόνια στην Ιδεολογική λεκάνη ε, της περιοχής Ρονάλπ, Ροδανού Άλπαιων στη Γαλλία και έδειξε ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει διαφορά σε ό,τι την τιμή και την υπηρεσία μεταξύ δημόσιας διαχείρισης ή ιδιωτικής διαχείρισης. Το θέμα είναι οι υποδομές για μακρά χρονική περίοδο. Εκεί τι γίνεται. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να πλαισιωθούν οι συμβάσεις να ελέγχεται με σοβαρό τρόπο η παροχή των υπηρεσιών. Νομίζω ότι συμφωνούμε από αυτόν τον σημείο. Ευχαριστώ. Thank you very much. And now, Madam Switza. Ευχαριστώ, κυρία Σουίτσα. Ευχαριστώ την εισηγήτρια. Ε, είναι αυτή η πρώτη δημόσια συζήτηση και θέλω να πω και εγώ δύο λόγια. Αν κάνουμε δημοψήφισμα για αυτό το θέμα, το αποτέλεσμα θα ήταν 95% όπως συνέβη πρόσφατα στην Ιταλία. Γιατί το θέμα έχει τεράστια σημασία και νομίζω ότι και το νερό σαφώς δεν είναι εμπόρευμα, είναι δημόσιο αγαθό. Ούτε μπορούμε να βλέπουμε ως ε, εμπορικό ε, προϊόν το νερό. Ο αριθμός πάνω από 1,5 εκατομμύριο υπογραφών δείχνει πόσο οι Ευρωπαίοι πολίτες νιώθουν για το ζήτημα αυτό. Οι υπογράφοντες ε, ζητούν τρία πράγματα που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά και τα θεσμικά όργανα μαζί με τα κράτη-μέλη πρέπει να επιτρέψουν, να διασφαλίσουν σε κάθε πολίτη το δικαίωμα πρόσβαση σε νερό και αποχέτευση. Επίσης πιστεύω ότι η υδάτινη πόρη, όπως αναφέρεται και στο σημείο 2, δεν πρέπει να υπόκεινται σε κανόνες της εσωτερικής αγοράς και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να μας βοηθήσει ε, σε σχέση με την ελευθέρωση. Πρέπει να ε, κάνουμε πιο πολλές προσπάθειες όλοι μας, ιδιαίτερα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο ε, σε, και σε επίπεδο κρατών μελών και σε ενωσιακό επίπεδο, το ώστε το καθολικό δικαίωμα πρόσβαση στο νερό να κατοχυρωθεί για όλους και περιμένω τη συνέχεια που θα δοθεί σε αυτή την ε, Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Ελπίζω να πετύχουν. Όταν μιλάμε για αναπτυσσόμενες χώρες έχουν πολλά προβλήματα πραγματικά και πρέπει να υποστηριχθούν με ενωσιακά κονδύλια ούτω ώστε όλοι οι πολίτες του πλανήτη να έχουν πρόσβαση στο νερό. Τέλος, για να κλείσω, αν ε, το νερό έπαιζε περισσότερο ρόλο στις διεθνείς σχέσεις ε, όπως έγινε με το πετρέλαιο είμαι βεβαία ότι η πρωτοβουλία μας θα ήταν πιο ευπρόσδεκτη. Όμως δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον. Στην Κροατία, την πατρίδα μου, που είναι η τρίτη χώρα σε υδάτινους πόρους μετά την Νορβηγία και την Ισλανδία. Γνωρίζουμε πολύ καλά τη σημασία του πόρου αυτού. Γι' αυτό είμαι υπέρ της πρωτοβουλίας και ελπίζω ότι μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το εθνικό, το περιφερειακό και το τοπικό επίπεδο θα μπορέσουμε να βρούμε μια λύση. Τώρα, για τις σε ιδιωτικού δημοσίου τομέα, νομίζω ότι ε, είναι ευπρόσδεκτες, αλλά οι συμβάσεις για τις παραχωρήσεις είναι πολύ σημαντικές και πρέπει να δούμε ε, πώς θα γίνει η διαχείριση του ύδατος. Ευχαριστώ. Τελευταίος που θα πάρει το λόγο και μετά ο κύριος Τούρμες θα είναι ο τελευταίος. Ευχαριστώ. Καθυστέρησα γιατί είχαμε ψηφοφορία στην Ήτρα και πήρε πιο πολύ χρόνο. Συνάδελφοι, το νερό είναι ζωή. Χωρίς νερό δεν υπάρχει ζωή. Και γι' αυτό πρέπει να δούμε την εμπλοκή των πολιτών που ανησυχούν για το νερό και τη διαχείρισή του ε, που μας παρακολουθούν σχετικά με το τι κάνουμε για το νερό αυτό πρέπει να το δούμε ως ευκαιρία ε, ευαισθητοποίησης η πρωτοβουλία για το νερό ήταν η πρώτη, δηλαδή είναι ιστορική ε, πρωτοβουλία και ιστορικό επίτευγμα των πολιτών στην Ευρώπη με αντικείμενο το νερό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προσέφερε ελάχιστες υπηρεσίες θα έλεγα μάλλον ενοχλούνται που, από τους πολίτες που δραστηριοποιούνται παρά χαίρονται. Δεν είναι καλό αυτό. Εμείς πρέπει να είμαστε ευτυχείς για το γεγονός ότι δείχνουν ενδιαφέρον για αυτό που κάνουν οι πολίτες. Το νερό είναι ζωή λοιπόν, πάνω απ' όλα και αυτό είναι πολύ σημαντικό ιδιαίτερα στις τρίτες χώρες και γι' αυτό είναι καλό στην έκθεσή μας να τονίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει περισσότερα από ό,τι κάνει μέχρι τώρα για να βοηθήσει όλους τους πολίτες, τα παιδιά, τις γυναίκες, σε όλο τον κόσμο για να έχουν όλοι πρόσβαση στο νερό. Το άλλο θέμα είναι το νερό στην Ευρώπη. Ε, στην Ήπειρό μας οι περισσότεροι ε, άνθρωποι έχουν πρόσβαση στο νερό μια κοινότητα όμως καμιά φορά δεν έχει πρόσβαση που είναι οι κοινότητε των Ρωμά και πρέπει αυτό να το υπογραμμίσουμε και να μην ε, κάνουμε παρελκυστική τακτική. Πρέπει να έχουν και αυτή πρόσβαση στο νερό. Τώρα, ένα μεγάλο θέμα είναι η σύμβαση για τις παραχωρήσεις. Εκεί θα δοθεί μάχη. Νομίζω ότι πρέπει να μην επιτρέψουμε ε, παιχνίδια να κάνει Κομισιόν. Ε, η πλειοψηφία ήταν πολύ μεγάλη στο Κοινοβούλιο και είπε ότι δεν πρέπει να ε, ξανανοίξει η συζήτηση για τις παραχωρήσεις λόγω της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας των Πολιτών. Ε, το νερό είναι πολύ κοντά στο δημόσιο συμφέρον και δεν βλέπω να έχει συμφέρον η Ευρωπαϊκή Ένωση να δίνει μάχη για την ιδιωτικοποίηση ε, στο νερό. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να το αποδεχτεί η Κομισιόν. Θα πρέπει όσο γίνεται περισσότερο να μείνει στα χέρια του δημοσίου. Βέβαια, ε, ε, σε κάποιες υπηρεσίες, για κάποιες υπηρεσίες μπορεί να υπάρξουν και ιδιωτικές εταιρείες. Η ποιότητα του νερού πρέπει να τονιστεί περισσότερο. Υπάρχει μια πρόσφατη μελέτη από ένα γερμανικό πανεπιστήμιο το οποίο για πρώτη φορά έσκαψε λίγο περισσότερο στο θέμα των ζυζανιοκτώνων, παρασιτοκτώνων και κατέληξαν ότι περίπου το 40% των δειγμάτων παρουσιάζουν κατάλοιπα. Ε, είναι πολύ δαπανηρό να αφαιρεθούν αυτά τα κατάλοιπα από το πόσιμο νερό. Οπότε η σύγκρουση που έχουμε και μια αντίφαση δεκαετιών που δεν μας έχει απασχολήσει όπως θα έπρεπε είναι αφενός η χρήση των ζυζανιοκτώνων παρασυντοκτώνων και οι πολύ για πραγματικά βλαβερές επιπτώσεις του στο πόσιμο νερό. Στις εκθέσεις μας πρέπει να είμαστε πιο σαφείς πάνω σε αυτό. Αν θέλουμε το νερό να είναι πόσιμο, το, το νερό της βρύσης, που θα έπρεπε να μπορούμε να το πίνουμε γιατί είναι πιο φθηνό Και όταν μιλάμε για την κυκλική οικονομία ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την ανακύκλωση, τα πλαστικά μπουκάλια κλπ. Δηλαδή εδώ πέρα στο κοινοβούλιο ε, έχουν γίνει κανόνα τα πλαστικά μπουκάλια για το νερό. Ενώ στην Ευρώπη έχουμε τη δυνατότητα να πίνουμε καλό νερό από τη βρύση και θα πρέπει στην έκθεσή μας να το τονίσουμε ότι θέλουμε το νερό αυτό να το πίνει ο κόσμος ώστε να μην ε, ε, ξακοντίζεται τεχνητά η κατανάλωση ε, του νερού. Ε, ε, νομίζω ότι χρειάζεται μεγαλύτερη συνέπεια πολλές φορές. Υπάρχει ε, η αίθουσα όπου συνεδριάζει η ομάδα των Πρασίνων και εκεί ε, είπαμε ότι πρέπει να υπάρχει βρύση και το κάναμε αυτό ε, και ε, ίσως πρέπει να το κάνουμε και σε άλλες αίθουσες για να γλιτώσουμε από τη σκλαβιά του πλαστικού μπουκαλιού. Ευχαριστώ. Δύο ακόμη συνάδελφοι ζήτησαν το λόγο, ο κύριος Φλάναγκαν. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν να συγχαρώ την συνάδελφο Μπόιλεν για την εξαιρετική δουλειά. Το νερό είναι πολύ σημαντικό και η παροχή του, αλλά και αυτό έχει να κάνει και με την αξιοπιστία των ε, Ευρωπαϊκών Πρωτοβουλειών Πολιτών. Δεν ξέρω πόσο σοβαρά λαμβάνεται η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Όταν ε, ε, ε, οι πολίτες αμφισβητούν ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση. τώρα με την πρωτοβουλία θα εισακοστούν. δηλαδή πολλές φορές δίνουμε ελπίδα στον κόσμο ότι δήθεν έχουν ένα λόγο, ενώ στην πραγματικότητα δεν εισακούονται. Είναι ενδιαφέρον αυτό που λένε κάποιοι ορισμένοι ότι η Κομισιόν δεν έχει αρμοδιότητα να αποφασίσει αν έχουμε δικαίωμα για νερό κλπ γιατί αυτό είναι στα κράτη, θέμα κρατών μελών. Στην ε, χώρα μου, στην Ιρλανδία, το 2010 όταν αναγκαστήκαμε να διασώσουμε μη συστημικές ε, τράπεζες πληρώντας δεκάδες δις ευρώ, όχι μόνο αναγκαστήκαμε να το κάνουμε αυτό, ε, μετά από επιστολή του Jean-Claude Trichet, ε, ε, τον τέλειο gentleman, το λέω λίγο ειρωνικά, ε, εκεί ε, ο κύριος Τρισέ είχε πει ότι οι κυβερνήσεις και αυτό πρότεινε δηλαδή για το 2012 και το 2013 όταν εμείς ε, είχαμε αυτό το πρόβλημα θα έπρεπε να είχε κάνει αξιολόγηση η κυβέρνηση σχετικά με τις, ε, υπο, τις, ε, ε, τους οργανισμούς ίδρευσης, οι εταιρείες ίδρευσης, ούτως ώστε να αρχίσουν το 2012-2013 να αρχίζουν να επιβάλλουν χρέωση για το νερό με, μεγαλύτερη. Τώρα μας λέγουν ότι δεν έχουν αρμοδιότητες, ενώ παλαιότερα ο εκπρόσωπος των, τρα, των τραπεζών σε αυτήν την υποτιθέμενη ένωση που λέγεται κοινότητα ήρθε και μας είπε τι έπρεπε να κάνουμε με το νερό. Ε, είναι υποκρισία. Όταν ε, ταιριάζει στα συμφέροντα των μεγάλων μπορεί να γίνει, όταν, είναι, ε, όταν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μικρών δεν μπορεί να γίνει. Θα πρέπει να αρχίσουμε να κοιτάμε τα συμφέροντα του μικρού ανθρώπου, των απλών ανθρώπων. Εγώ άρχισα ως υπέρμαχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τώρα την απεχθάνομαι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ε, λέει κυρία Πετήρ. Αυτή η πρωτοβουλία που υποστηρίζεται από 1,6 εκατομμύρια ανθρώπους είναι σημαντική διότι το νερό είναι ζωτικό δημόσιο αγαθό. Ε, φιστώ την προσοχή σας σε ορισμένα θέματα. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι κάποιοι πτωχοί άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση στο νερό Ζητώ λοιπόν να δημιουργηθεί ε, ένα κοινωνικά ε, ελάχιστο ε, όριο κατανάλωσης. Είναι λυπηρό ότι ιδιωτικοποιείται η διαχείριση του ύδατος, των υδάτων. Αυτό είναι τελείως αντιδημοκρατικό. Είναι σημαντικό να θεσπίσουμε μηχανισμούς κατά της υπερβολικής ιδιωτικοποίησης των υδάτων και την ανεξέλεγκτη ε, εκμετάλλευση επίσης της άμμου και των χαλικιών. Δεν υπάρχει σαφής ε, ε, στρατηγική για την εξαγωγή υδάτων. Και αυτό πρέπει να το δούμε και να το αντιμετωπίσουμε. Διότι έτσι, αλλιώς θα ανοίξει ο δρόμος για, τους, για τις πολυεθνικές και οι μάνατζερ θα κοιτάξουν να αποκομίσουν κέρδη ε, σε βάρος ε, ενός πολύτιμου αγαθού που δεν ανανεώνεται. Ε, έχουμε πάρα πολλές συγκρούσεις που οφείλονται στη λειψιδρία. Το νερό, όπως είπαμε, είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα. Η πρόσβαση στο νερό και πρέπει να το διατηρήσουμε. Οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν το δικαίωμα να επηρεάζουν την λήψη αποφάσεων στον τομέα της διαχείρισης των υδάτων. Και είναι σημαντική η δημόσια παροχή ύδατος. Η Κροατία είναι η τρίτη, όπως ελέγχθη, χώρα εις ό,τι αφορά την παροχή ποσίμου ύδατος. Και βέβαια είμαι υπέρ της διατήρησης των πηγών ύδατος από τη ρήπανση και την εκμετάλλευση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Και τώρα δίνω το λόγο στην Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είμαι από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Κομισιόν. Να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και όλους όσους συνεργάστηκαν για την προετοιμασία και παρενέβησαν σήμερα. Θέσατε πολλά και σημαντικά και κάποια επικριτικά είπατε, αλλά είναι ευπρόσδεκτα όλα στη συζήτηση για αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία. Θα παρακολουθούμε και θα δούμε τι συνέχεια θα δοθεί στην Ολομέλεια. Θέλω να κάνω τρεις παρατηρήσεις και να σας δώσω και κάποιες ε, χρήσιμες ίσως πληροφορίες για τη συνέχιση της συζήτηση και την τελική έκθεση. Πρώτον, για να απαντήσω. Στην ε, Κομισιόν αναγνωρίζεται σαφώς η σημασία του νερού ως δημόσιο αγαθό που είναι σημαντικό για τη διατήρηση της ζωής. Αυτό προκύπτει σαφώς από την ανακοίνωση και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκή Ένωση που συνεχώς έπαιζε θετικό ρόλο για να εξασφαλίζεται πόσιμο νερό για όλους και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός αυτής. Δεύτερον, θυμίζω ότι σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες ύδατος στην εσωτερική αγορά η απάντηση ε, διευκρινίζει την αρχή της ουδετερότητας. Ε, πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι ουδέτερη σε σχέση με τις εθνικές αποφάσεις σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, είτε είναι ιδιωτικό, είτε είναι δημόσιο, είτε είναι σε, ε, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Όλα αυτά εμείς τα χαιρετίζουμε στο βαθμό που βελτιώνουν τις υπηρεσίες ύδατος και την πρόσβαση των πολιτών σε αυτές. Τρίτον, ευχαριστώ τον Κλοντ Τούρμες Βλέπετε, δεν έχω πλαστικό μπουκαλάκι, ε, το κάνω refill, το ξαναγεμίζω το μπουκαλάκι μου. Ε, τους τελευταίους μήνες υπάρχουν κάποιες εξελίξεις, ίσως δεν ξέρετε, στις 20 Απριλίου η Επιτροπή πώς μου είδα τόσα ομόφωνα υποστήριξε την αναθεώρηση των ε, παρατημάτων 2 και 3 στην οδηγία πόσιμου νερού που εκτός από κάποια τεχνικά θέματα το σημαντικό είναι ε, αν δεν έχουν αντιρρήσει στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο στη διαδικασία ελέγχου, θα μπορούμε να κάνουμε περισσότερη παρακολούθηση των υδάτων και αυτό θα βελτιώσει και το ε, πρόβλημα παρακολούθησης ε, της παροχής περιορισμένων ποσοτήτων ύδατος γιατί υπάρχουν ε, κάποιοι που ε, αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Αυτά είναι πρόσφατες εξελίξεις. Τώρα αξιολογούμε ως άμεση επίπτωση της πρωτοβουλίας των πολιτών και είναι στο πρόγραμμα της δράσης της Κομισιόν την οδηγία που σήμου ε, ε, Έχουμε και ένα, μια ιστοσελίδα Safe to Drink, ασφαλές για να το πίνουμε. Στις 26 Μαΐου θα γίνουν και διαβουλεύσεις με τους δημόσιους εμπλεκομένους και είστε και εσείς προσκεκλημένοι. Τελευταίο, πολύ μιλήσατε για τη λήψη ιδρία, τα επιφανειακά ύδατα, τους ποταμούς, το πόσιμο ίζορ και πώς θα αντιμετωπίζουμε όλα αυτά. Τις τελευταίες εβδομάδες δημοσιεύτηκε μια αξιολόγηση για το πώς τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν την οδηγία πλαίσιο για το πόσιμο ίδωρ επιτόπου. Ε, 53% μπορεί να πει κανείς ε, να δει το ποτήρι μισοάδιο ή μισογεμάτο 53% ε, είναι η γεματο 53 ειναι η εφαρμογη με το οικολογικό καθεστώς και αυτό επηρεάζει σε τελευταία ανάλυση το πόσο πόσιμο νερό έχουν οι πολίτες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν προχωράει το θέμα Ακούσαμε πολλά σημαντικά σήμερα. Θα παρακολουθήσουμε με ενδιαφέρον τη συνέχεια και θα επανέλθουμε όταν η τελική έκθεση εγκριθεί από την Ολομέλεια του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα δώσω ξανά το λόγο ε, στην εισηγήτρια για να ολοκληρωθεί η συζήτηση. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους που συνέβαλαν στη σημερινή συζήτηση και προσπάθησα να σημειώσω όλα τα σχόλια και θα προσπαθήσω στην απάντησή μου να τα καλύψω. Πρώτα απ' όλα για την αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα ύδατα και τη διαχείρισή τους και την διοκτησία τους. Ναι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχώς διατείνεται ότι δεν έχει αρμοδιότητα, είναι κάτι που εξαρτάται από τα κράτη-μέλη. Αλλά και ο συνάδελφος από την Ιρλανδία είπε ότι οι δράσεις της είναι πολύ διαφορετικές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σαν μέρος της Τρόικα έχει υπονομεύσει τη δυνατότητα των κρατών μελών να αποφασίζουν το πώς θα διαχειρίζονται τα θέματα των υδάτων και της αποχέτευσης και ποιος είναι ιδιοκτήτης. Πρέπει να γνωρίσουμε ότι αυτή η έκθεση δεν λέει στα κράτη-μέλη τι θα πρέπει να κάνουμε το νερό του αλλά αυτό που θα έπρεπε να προστατεύσουμε την δυνατότητα επιλογή. Και αυτό είναι που υπονομεύεται από τι δράσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και εκτό τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, αυτό είναι πιο ξεκάθαρο όσον αφορά την αιρεσιμότητα τη ιδιωτικοποίηση που επιβάλλεται σε πολλά προγράμματα των απτυσσομένων χωρών. Και κάτι άλλο που ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία της πρωτοβουλίας πολιτών ήταν να βγει το νερό από τη διαδικασία παραχωρήσεων από βράση του Μισελ Μπαρνιέ και είναι ενδιαφέρον να βλέπουμε ότι αυτό αναθεωρείται. Συμφωνώ με αυτό που είπαν συνάδελφοι. Ελπίζω αυτή η έκθεση και η πρωτοβουλία των πολιτών να μην χρησιμοποιηθεί ως απόπειρα ε, να προωθηθεί η απελευθέρωση των υδάτων. Όσον αφορά το ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό, το Κοινοβούλιο δύο φορές και είναι σημαντικό αυτό, αναγνώρισε το νερό σαν ανθρώπινο δικαίωμα. Αναγνωρίζεται σαν εν, μοναδικό ε, δημόσιο αγαθό σε ένα ψήφισμα που πέρασε για την εσωτερική αγορά και είναι και κοινό πόρο το νερό για, τον, ε, το ανθρώπινο είδο και το νερό δεν πρέπει να υπόκειται στου κανόνε εσωτερική αγορά. Και η πρόσβαση στο πόσιμο νερό είναι ζωτικό θεμελιώδες δικαίωμα και δεν είναι οικονομικό εμπορεύσιμο προϊόν που υπόκειται στους κανόνες αγοράς και πέρασε και ένα ψήφισμα που αναφέρεται σαν ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό του 2006 στο τέταρτο φόρουμ, το Παγκόσμιο Φόρουμ για το νερό. Συμφωνώ όσον αφορά την οδηγία πλαίσια για το νερό ότι πρέπει να διαφυλάξουμε το νερό. Η οδηγία ως έχει δεν αναφέρεται στην εκπαίδευση, στην ενημέρωση και καμιά φορά οι πολίτες κατηγορούνται για τη σπατάλη του νερού. Ε, και εμείς κάνουμε παρόμοια πράγματα και αφήνουμε τις βρύσες να τρέχουν. Οι περισσότεροι άνθρωποι Ακόμα και στην Ιρλανδία που υπάρχει νερό άφθονο, ο κόσμος γνωρίζει ότι πρέπει να ε, μη σπαταλάνε το νερό και κατά μέσο όρο είναι υπεύθυνοι, αλλά θα πρέπει η εκπαίδευση να μπει στην οδηγία πλαίσια για το νερό. Μιλάμε για τη συντήρηση, για τη διαφύλαξη του νερού. Αλλά δεν χρειάζεται εκπαίδευση μόνο οι πολίτε, αλλά και η γεωργία και η βιομηχανία έχουν ρόλο να παίξουν. Χρησιμοποιούν περισσότερο νερό από ότι οι πολίτε. Όσον αφορά τη διαχείριση και τη δημόσια κυβέρνηση, ακούστηκαν πολλά σχόλια, καλό αυτό. Αναφέρθηκαν στην ανάγκη οι καταναλωτές και οι πολίτες να έχουν λόγο σχετικά με τη διαχείριση του νερού. Και ε, εδώ έχουμε περιθώρια στην έκθεση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιδιώξουμε εφαρμογή πολιτικής για τη συμμετοχή των πολιτών στη διαχείριση του νερού θα πρέπει να έχουν λόγο είτε απευθύνονται σε ιδιωτικό φορέα, δημόσιο φορέα διαχείριση των υδάτων, πρέπει να έχουν λόγο όσον αφορά τη διαχείριση των υδάτων, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό τον όρο την ύπαρξή του. Και μόνο μέσω δημόσια διαχείριση οι αποφάσει μπορούν να θεωρηθούν ω διαφανεί και τα μεγάλα έργα της υποδομής ε, ε, πρέπει να ε, υπόκειται στον έλεγχο και στην κρίση των πολιτών. Και θα πρέπει οι υπηρεσίες παροχής νερού να μην οδηγούν σε περιβολικά κέρδη για τους μετόχους. Σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσης βλέπουμε ότι το κόστος του νερού ανέβηκε πάρα πολύ, πολύ πάνω από το επίπεδο του πληθωρισμού και έχει φτάσει μέχρι το 6% του εισοδήματος των οικοκυριών. Λοιπόν, φθηνό νερό και πρόσβαση στο νερό είναι ένα αυξανόμενο πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να καλυφθεί είτε μέσω κανονισμού είτε μέσω δημόσιας διαχείρισης. Ο συνάδελφος FT αναφέρθηκε στην ποσόστοση και αναφέρθηκα στον ε, την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας που θεωρεί ότι είναι ανάμεσα στα 50 με 100 λίτρα νερού την ημέρα που ε, απαιτούνται για την κάλυψη βασικών αναγκών. Εγώ ξεκίνησα, μάλλον μπορούμε να συζητήσουμε την ποσότητα, αλλά συμφωνούμε ότι υπάρχει ελάχιστη ποσότητα νερού που είναι θεμελιώδης για την ανθρώπινη ζωή. Αναφέρθηκε ένα είδος βαθμολόγησης. Αν η βαθμολόγηση αφορά συγκρίση η σύγκριση, τη διαχείριση των υδάτων πρέπει να παρέχεται κοινωνική προστασία, να συμπεριλαμβάνεται κοινωνική προστασία. Είναι διαφορετικό αγαθό, πρέπει να προστατεύεται. Ε, δεν θα πρέπει η διαχείριση να βασίζεται μόνο σε οικονομικές ή χρηματοπιστωτικές πτυχές. Τόσον αφορά τι συμπράξει του δημόσιου τομέα και δημόσιου ιδιωτικού τομέα, Αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία των πολιτών Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να αναλύσουμε περαιτέρω το θέμα και να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ούτω ώστε να προωθήσουμε αυτή τη μορφή συμπράξεων και κυρίω με την υποστήριξη των δημοσ... συμπράξεων του δημόσιου τομέα που έτσι μπορούν να βοηθήσουν τι αναπτυσσόμενε χώρε να βελτιώσουν την ποιότητα του νερού και να γίνει πόσιμο. Και τέλο κάτι άλλο σαν αφορά την πρωτοβουλία των πολιτών. Αυτή καθ' αυτή διάβασα διάφορες εκθέσεις θέσεις μετά την πρώτη πρωτοβουλία των πολιτών. Είναι σημαντικό ότι το δικαίωμα στο νερό είναι η πρώτη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών που ενεκρίθη που ξεπέρασε την ποσόστοση του ενός εκατομμυρίου υπογραφών και θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι σε αυτή τη φάση οι πολίτες εμπιστεύονται τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ή μάλλον η εμπιστοσύνη τους είναι πολύ χαμηλή όσον αφορά τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Τους προσφέραμε αυτή τη δημοκρατική διαδικασία στη Λισαβόνα, θεωρούσα ότι ήταν ασθενής τότε την έχουμε τώρα και αν αποδυναμώσουμε αυτό το εργαλείο περαιτέρω με πολύ ε, κακές αντιδράσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό θα είναι πάρα πολύ επιβλαβές για την ε, δημοκρατία. Και σταματώ εδώ Πρόεδρε λέγοντας αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα έχουμε μόνο άλλο ένα σημείο. Α, προθεσμίες για την υποβολή τροπολογιών 21 Μαΐου. Ψηφοφορία. επιτοπή ΕΝΒΙ 25 Μαΐου. Στην Ολομέλεια θα ψηφίσουμε τον μήνα Σεπτέμβριο. Μόνο άλλο ένα σημείο έχουμε στην ημερήσια διάταξη. Περιμένουμε όμως για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προτείνω διακοπή 5 λεπτών για να περιμένουμε για τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μετά συνεχίζουμε. Thank you Okay, I think that the Commission is arrived and then uh, we... Νομίζω ότι κατέφτασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορούμε να ξεκινήσουμε ξανά τη συνεδρίαση μας. Το σημείο 19α λοιπόν. Ε, Κατεξοδότηση στην πράξη για εξαίρεση για το κάδμιο σε διάφορα φωτιστικά ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεχθήκαμε αίτημα των Πρασίνων επ' αυτού. Ας μας εξηγήσει τα πράγματα ο κύριος Τέιλορ. Εν ονόματι της ομάδας των Πρασίνων. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα γνωρίζετε ίσως ότι μέλος των Πρασίνων η Jill Evans ήταν η για την αναδιατύπωση της οδηγίας για τον περιορισμό επικινδύνων ουσιών στον ηλεκτρονικό και ηλεκτρικό εξοπλισμό. Η οδηγία ΡΟΣ, όπως ονομαζόταν, 2011. Μας ενδιαφέρει η πλήρης και σωστή εφαρμογή της ανλογοδηγίας. Περιορίζει η οδηγία τη χρήση κάποιων επικινδύνων ουσιών. Όχι μόνο για να η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, αλλά και για να συμβάλλουμε στην περιβαλλοντική ανακύκλωση των αποβλήτων από πλευράς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Και στην τελική σκέψη 8 της οδηγίας λέει ότι ο περισμός της χρήσεως των εν λόγω επικινδύνων ουσιών πιθανότατα θα αυξήσει τις δυνατότητες που υπάρχουν και το οικονομικό κέρδος της ανακύκλωσης αποβλήτων. Αποβλήτων που προέρχεται από ηλεκτρονικό και ηλεκτρικό εξοπλισμό. Έτσι, η σωστή εφαρμογή της οδηγίας αυτής είναι κρίσιμο στοιχείο στην κουβέντα που γίνεται τώρα για την κυκλική οικονομία. Έχει δικαίωμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θετήσει εξαιρέσει υπό τη μορφή κατεξουσιοδότηση πράξεων υπό τους όρους που παρατίθενται στο άρθρο 5. Στην κατεξουσιοδότηση πράξη που έχουμε μπροστά μας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει επέκταση παρέκκλησης που υπάρχει για τη χρήση καδμίου στις, τα LEDs για τις οθόνες και για τους λαμπτήρες και να χρησιμοποιηθεί το κάδμιο που έχει ε, κοιλίδες ε, ε, κλαντικές και συγκεκριμένες εξαιρέσεις για το κάδμιο περιέχει αυτές τις τις, ε, τις κουκίδες η κατάσταση εδώ διαφέρει σχέση με την ΡΟΣ, με την οδηγία αυτή την παλιά που εφητήθηκε για να αντικατασταθούν οι χρήσει κάποιων επικινδύνων ουσιών όποτε αυτό είναι δυνατόν. Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχουν ε, προϊόντα που χρησιμοποιούν ε, καδμίου με, ε, κουκίδες, καδμίου, με κουκίδες καδμίου στην αγορά και δεν χρησιμοποιείται στις οθόνες. Άρα δεν τίθεται θέμα να απαλλαγούμε από το κάδμιο σε υφιστάμενες συσκευές, αλλά κατά πόσο θα επιτρέψουν στο κάδμιο να χρησιμοποιηθεί σε νέες εφαρμογές και συσκευές, διότι είναι πολύ τοξικές οι ιδιότητες του. Αλλά η χρήση στις συσκευές ίσως τελικά να είναι υποφελής όσον αφορά το περιβάλλον και όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια. Η οδηγία λοιπόν θα επέτρεπε εξαίρεση, αλλά μόνο αν αυτό που αντικαθιστά το κάδμιο δεν είναι πρακτικός εφαρμοστή είτε υποκατάστατα του καδμίου δεν ήταν αξιόπιστα ή υποκατάστατα είχαν περισσότερες αρνητικές συνέπειες από ό,τι θετικές. Ας δούμε ένα-ένα τα στοιχεία αυτά. Οι συνθήκες πληρούνται για τους λαμπτήρες που περιέχουν κάδμιο που περιέχει κβαντικές κουκίδες. Η απάντηση είναι όχι διότι τέτοια προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα ακόμα. Και όπως αναγνωρίζει η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οσδήποτε θετικός αντίκτυπος στο περιβάλλον δεν μπορεί να αποδειχτεί, είναι θεωρητικός, υποθετικός. Γι' αυτό οι σύμβουλοι που προσέλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέστησε να μην συνεχιστεί η εξαίρεση για τους λαμπτήρες. Δεύτερον, πληρούνται οι όροι για τις οθόνες που περιέχουν κάδμιο με κβαντικές κουκίδες. Η απάντηση είναι ουχή, διότι το κάδμιο με κβαντικές κουκίδες είναι διαθέσιμο τεχνικά. Μπορείς να βρεις τηλεοράσεις που περιέχει αυτή την ουσία και στο Βέλγιο και στο Ηνωμένο Βασίλειο τηλεοράσεις με αυτό το στοιχείο. Αυτό δεν ίσχυε πριν από ένα χρόνο. Το Ινστιτούτο Όκο έκανε αξιολόγηση και είπε ότι έπρεπε να προβλέπεται συγκεκριμένη εξαίρεση για τρία χρόνια. Πολλά συνέβησαν έκτοτε, τον τελευταίο χρόνο. Γι' αυτό ως νομοθέτες πρέπει να είμαστε ενήμεροι και σύγχρονοι. Μη θεωρείτε σας παρακαλώ ότι επικρίνουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται κάποια δεδομένη χρονική στιγμή και αλλάζουν τα πράγματα μετά. Όμως θα καταλαβαίνετε κι εσείς ότι εμείς στο Κοινοβούλιο πρέπει τουλάχιστον να προσπαθούμε να παίρνουμε αποφάσεις υπό το φως της παρούσης καταστάσεως και ουχή της προηγουμένης. Μπορείτε να πείτε ότι δεν αρκεί αυτό. Ότι υπάρχει υποκατάστατο που βασίζεται διαφορετική ουσία και ότι η χρήση της αναλλακτικής ουσίας είναι πλέον υποφελής τα φωσφορούχα διάφορα δεν είναι θετικά και ίσως να αντικατασταθούν. Όμως δεν περιορίζονται ακόμα. Και είναι σε καλύτερη θέση από το κάδμιο. Λοιπόν, οι οθόνες που έχουν κβαντικές κουκίδες που δεν έχουν κάδμιο ε, έχουν ίση κατανάλωση ενέργειας και ίδιες ιδιότητε ιδιότητες απεικόνησης δεν υπάρχουν ε, περιβαλλοντικά ωφέλη για να χρησιμοποιήσουμε κάδμιο με ε, κβαντικές κουκίδες έναντι ε, ουσίας που δεν περιέχει ε, κάδμιο. Άρα έχουμε εναλλακτικές ασφαλέστερες. Άρα δεν υπάρχει λόγος να προβλέψουμε εξαίρεση για το κάδμιο με κβαντικές κουκίδες στις οθόνες, αφού υπάρχουν άλλες λύσεις. Άρα, έχω τρεις ερωτήσεις για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτα, γιατί θέλετε να δώσετε παρέκκληση στο κάδμιο που περιέχει κβαντικές κουκίδες στις, στους λαμπτήρες LED παρά τις συστάσεις του συμβούλου σας και δοθέντος ότι αδίποτε περιβαλλοντικά ωφέλη αυτών των λαμπτήρων εν συγκρίση με, τις, με τους συμβατικούς λαμπτήρες δεν έχουν αποδειχθεί. Δεύτερον, δοθέντων των προσφάτων εξελίξεων όσον αφορά την χρήση των κουκίδων χωρίς κάδμιο με παρόμοια ή καλύτερη απόδοση ενεργειακή και απεικόνιση χρωμάτων όπως το κάδμιο με κβαντικές κουκίδες. Θεωρείτε λοιπόν ότι η δικαιολόγησή σας Όταν διατείνεστε ότι ε, οι κουκίδες, οι κβαντικές κουκίδες χωρίς κάδμιο δεν είναι διαθέσιμες, αυτό διατείνεστε, όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν, εξακολουθεί να ισχύει. Και θέλετε να δώσετε διπλή εξαίρεση για την εξαίρεση για το κάδμιο με κβαντικές κουκίδες σε δύο επίπεδα, σε υψηλότερο και χαμηλότερο. Πώς δεν συνδέονται οι δύο εξαιρέσεις στα δύο επίπεδα. Η ειδικοί εξαίρεση με χαμηλότερο επίπεδο ισχύει όταν η γενική με τα υψηλότερα επίπεδα περιεκτικότητας έχει εκπνεύσει. Λοιπόν, περιμένω πώς και πώς να ακούσω τις απαντήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Μπέρντερ για άλλη συμπληρωματική ερώτηση και μετά θα δώσουμε το λόγο στην Κομισιόν για να απαντήσει. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και το συνάδελφό μου, τον Γκίφ, που περιέγραψε σωστά τη θέση. Έχουμε μπερδευτεί όσον αφορά την παράταση της χρήσης του καδμίου. Είναι άκρος τοξική ουσία. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί χρειάζεται η παράταση αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βασίστηκε σε μελέτη του Ινστιτούτου ΟΚΟ, που είπε ότι η τεχνολογία ανευκαδμίου θα αργήσει να παραχθεί. Δεν ισχύει αυτό τώρα όμως. Σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος. Οι εταιρείε, κυρίως η Samsung, που ήδη έχει διαθέσει τηλεόραση στην αγορά και η LG φέτος, έκαναν τεράστιες επενδύσεις για να συμμορφωθούν με την εξάλληψη του καδμίου. Και κάποιες εταιρείε ήδη ανακοίνωσαν ότι έχουν και άλλες τεχνολογίες άνευ καδμίου. Οι ερωτήσεις μου. Τι μηνύματα στέλνουμε στις εταιρείε όταν θα τους δίνουμε περισσότερο χρόνο όταν λέγαμε πριν ότι θα πρέπει να κινηθούν, να απαλλαχθούν από την ουσία. Είναι πιο τοξική και από τον υδράργυρο. Και αυτή η επέκταση, αυτή η παράταση της παράκλη, παρέκκλησης πώς βοηθά την ευρωπαϊκή καινοτομία Πώς βοηθάει τη δημιουργία πρασίνων θέσεων εργασίας. Αυτή η παράταση θα ανοίξει την πόρτα σε φθηνότερες κινέζικες εισαγωγές. Και όλη η προσπάθεια που καταβάλαμε για την προώθηση πράσινων τεχνολογίας ποια ήτανε. Θέλαμε όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο να μειώσουμε τη χρήση των τοξικών ουσιών. Άλλη ερώτηση. Είδα εκτιμήσεις ότι η περίοδος της παράτασης σημαίνει ότι θα έχουμε 5 τόνους παραπάνω καδμίου που θα απελευθερωθεί στο περιβάλλον. Τι θα γίνει στο τέλος της ζωής των συσκευών, παραμένει στο περιβάλλον, απορροφάται πολύ γρήγορα από τα φυτά και τα φυλαστικά και από τους ανθρώπους. Ας το ξανασκεφτούμε, αυτό ζητάω. Δεν είναι μόνο το ζητάει το Κοινοβούλιο, αλλά και η χώρα μου, το Ηνωμένο Βασίλειο ε, και άλλες χώρες στο Συμβούλιο ανησυχούν πολύ και θα ήθελα να ακούσω ποιες είναι οι δικαιολογίες που έχει να μας δώσει το Συμβούλιο γι' αυτό και οι θέσει των χωρών στο Συμβούλιο δίνω στον κύριο Χούλιο Γκαρσία Μπόργες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το λόγο για να δώσει απαντήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να ζητήσω καταρχάς συγγνώμη για την καθυστέρηση. Απλά μας είχαν πει ότι η συζήτηση θα ξεκινούσε λίγο αργότερα. Πάντως είμαστε εδώ, ευτυχώς. Θα ήθελα καταρχάς να πω ότι πίσω από αυτή την κατεξουσιοδότηση πράξη υπάρχει πολύ, πολύ δουλειά. Αντικείμενο της ε, πράξης αυτής ε, είναι η εξαίρεση να παραταθεί για τις ε, συσκευές ε, φωτισμού και τις, ε, τους λαμπτήρες με κάδμιο. Δεκέμβριο του 2012 και Μάιο του 2013 έγινε μια διαδικασία που ακολουθήθηκε από διαδικασία διαβούλευσης, ολοκληρώθηκε έκθεση τον Απρίλιο του 2014. Το επόμενο βήμα ήταν η διαδικασία διαβούλευση ε, στην ομάδα εμπειρογνωμών, όπου η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτυχε ομόφωνη υποστήριξης. Και αυτό είναι σημαντικό ότι υπήρξε ομόφωνη υποστήριξη όταν έγινε διαβούλευση πέρυσι τον Ιούνιο. Δεν υπήρχε κανένας φορέας ε, που να θεωρεί ότι η εξαίρεση δεν ήταν δικαιολογημένη. Έπειτα είχαμε υπηρεσιακές διαβουλεύσεις και εγκρίθηκε η σχετική κατεξοδότηση η πράξη η οποία κοινοποιήθηκε δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα υπήρξε όμως ένα διαδικαστικό ζήτημα με τις ε, μεταφράσεις και κοινοποιήθηκε εκ νέου τελικά αυτή η πράξη το Συμβούλιο δεν ε, είναι αντίθετο. Ένα κράτος μέλος βέβαια έκανε μια πρόταση. Το έβαλε ένσταση. Πριν από δύο εβδομάδες συζητήθηκε στο Συμβούλιο αυτή η ένσταση. Και μόνο δύο ήταν υπέρ της ε, έστασης σε αυτή την πρόταση της Κομισιόν. Η περισσότερη συντριπτική πλειοψηφία υποστήριξε την εξαίρεση. Έρχομαι τώρα στην ουσία. Το περιεχόμενο. What is foreseen is to extend... Ε, αυτής πράξης προβλέπει την παράταση της ε, εξαίρεση 39 στο παράρτημα 3 του, της οδηγίας ΡΟΣ μέχρι το 2017 θα έπρεπε να έχει εκπνεύσει την 1η Ιουλίου του 2014 η εξαίρεση αυτή επειδή όμως υποβλήθηκε αίτημα για παράταση και αιτιολογήθηκε η παράταση, η διατήρηση της εξαίρεσης αυτής, θα έπρεπε να αξιολογηθεί αυτό το αίτημα. Προτείνουμε λοιπόν τώρα μια νέα εξαίρεση 39 Β, B για οθόνες που έχουν κουκίδες ε, κοβατικές με κάδμιο. Μια νέα εξαίρεση λοιπόν η οποία θα έχει πάρα πολύ αυστηρά κατόφλι πάνω από 2 νανογραμμάρια ένα τετραγωνικό μέτρο και θα ισχύσει μόνο μέχρι τον Ιούνιο του 2018. Η παράταση ισχύω της εξαίρεσης, της ισχύωσας εξαίρεσης, δεν φαίνεται να είναι επίμαχη. Είναι γεγονός ότι ο σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξέφρασε την άποψη ότι η εξαίρεση αυτή σε σχέση τι συσκευέ φωτισμού δεν εκπλήρωνε κάποιο σκοπό αφού δεν υπήρχε κάποια τέτοια συσκευή στην αγορά. Όμως, εξαίρεση αυτή περιλαμβάνεται στην οδηγία Ρώση σήμερα και υπήρξε άμεση αντίδραση των ε, φορέων οι οποίοι υποστήριζαν ότι γίνονταν εργασίες για την ε, παρασκευή μιας τέτοιας ε, συσκευής φωτισμού. Και ότι και αυτό θα έπρεπε να παραταθεί διάρκεια ίσως αυτής εξαίρεσης. Σίγουρα υπάρχει ένα θέμα αμφιλεγόμενο που είναι η νέα εξαίρεση 39B. Τη χρήση καρτμίου δηλαδή στη... με εκβατικές κουκίδες στις οθόνες. Για αυτό το θέμα. Θέλω να σας πω ότι του παρόντος και νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικότερο στοιχείο δεν υπάρχουν εφαρμογές ή συσκευές με εκβατικές κουκίδες που να είναι απαλλαγμένες από κάδμιο. Πράγματι πριν από ένα χρόνο. Οπότε και έγινε η αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι τεχνολογίες αναφικαδομίου δεν ήταν διαθέσιμες. Τώρα έχει πέρασει ένας χρόνος και φαίνεται ότι οι εναλλακτικές αυτές τεχνολογίες που είναι απαλλαγμένες από κάδμιο ίσως να διατεθούν τους επόμενους ε, μήνες. Πρώτα στην Κορέα και μετά στην Ευρώπη. Από μόνο του αυτό όμως δεν είναι ένας έγκυρος λόγος για την αντίθεση στην παράταση εξαίρεσης. Δεν υπάρχει ακόμη αυτή η τεχνολογία απαλλαγμένη, ε, πώς το λένε, άνευ καδμίου. Πουθενά δεν θα βρείτε ε, σε κανένα ράφι κανένας καταστήματος κάτι τέτοιο. Δεύτερον, η κατάργηση της εξαίρεσης ίσως δημιουργήσει κάποιες τρευλώσεις ε, της αγοράς ε, και πρόβλημα στην, στον εφοδιασμό. Γιατί δεν ξέρουμε κατά πόσον οι παρασκευαστές μπορούν να προμηθεύσουν την αγορά με αυτή την τεχνολογία ανευκαδμίου. Και το σημαντικότερο, οι εναλλακτικές, απαλλαγμένες από κάδμε τεχνολογίες δεν έχουν ακόμη καν δοκιμαστεί και αξιολογηθεί. διότι έχουν ε, χρήση φωσφορικών αλάτων του Ινδίου που και αυτό είναι, και αυτά είναι επικίνδυνο Θέλω να σας ε, παρουσιάσω ένα πρακτικό επιχείρημα που είναι σημαντικό και πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Εάν εκφράσει αντίρρηση το κοινοβούλιο θα πρέπει να ξεκινήσουμε ξανά από το μηδέν. Δηλαδή να επαναδρομολογήσουμε μια διαδικασία ε, που θα συνεπάγεται νέα επιστημονική αξιολόγηση, διαβουλεύσεις με την ομάδα εμπειρογνωμόνων, διυπηρεσιακές διαβουλεύσεις και όλα αυτά μπορεί να κρατήσουν δύο χρόνια και παραπάνω. Αυτό λοιπόν θα μας φέρει πολύ κοντά και στην ε, ημερομηνία λήξη της ισχύως αυτής της εξαίρεσης με βάση την ε, σημερινή, μάλλον την κατεξόδηση πράξη. Και η ισχύουσα εξαίρεση παραμένει σε ισχύ από τη στιγμή που έχουν υπάρξει αιτήματα παράτασης. Νομίζω ότι απάντησα τα περισσότερα από τα ερωτήματα που ετέθησαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί δηλαδή προτώνουμε αυτήν την εξαίρεση. Πολύ απλά παραλαμβάνω γιατί δεν είναι διαθέσιμες εναλλακτικέ τεχνολογίες αν ευκαδμίου ακόμη. Γιατί έχουμε αυτή τη διπλή εξαίρεση 39A και 39B. Η 39A είναι η ισχύουσα σήμερα εξαίρεση που περαβάνεται στην οδηγία ΡΟΣ και με τη νέα εξαίρεση για τις ακροβατικές κουκίδες στις οθόνες βάζουμε πιο αυστηρούς όρους για την εφαρμογή αυτής της εξαίρεσης. Και τώρα πώς αυτές οι δύο εξαιρέσεις αλληλοσυνδέονται μεταξύ τους, ε, η απάντηση είναι η εξής. Στην πρώτη περίπτωση έχουμε νωρίτερη ημερομηνία εκπνοής, ε, λήξης, ενώ για τις κβαντικές κουκίδες άνευ καδμίου στις οθόνες η εξέρεξη θα ισχύει για έναν ακόμη χρόνο. Ένα χρόνο παραπάνω σε σχέση με την πρώτη εξαίρεση, άρα θα μπορεί η αγορά να έχει το χρόνο στη διάθεσή της για να προσαρμοστεί στη νέα αυτή τεχνολογία. Και αν χρειαστεί θα έχουμε και τη δυνατότητα να ε, μελετήσουμε την αλλακτική τεχνολογία. Αν με επιτρέπετε τώρα να πω δύο λόγια γρήγορα γρήγορα για ένα επιχείρημα που ήδη αναφέρθηκε στη συζήτηση και συγκεκριμένα τις επιπτώσεις που θα έχει στην απασχόληση, στις θέσεις εργασίας. Κοιτάξτε, με βάση αυτά που γνωρίζουμε, η πρώτη εταιρεία η οποία θα αναπτύξει και θα διαθέσει το εμπόριο οθόνες ε, με κβαντικές κουκίδες ανευκαδμή, Δεν είναι ευρωπαϊκή εταιρεία. Άρα από αυτήν την έννοια, αυτό που ίσως κάνουμε είναι να άρουμε την, ε, αν άρουμε μάλλον την εξαίρεση, είναι να δημιουργήσουμε πιο ευνοϊκούς όρους και συνθήκες για εισαγωγές στην Ευρώπη. Για τις ε, εισαγωγές εκτονικών προϊόντων που παράγονται σε τρίτες χώρες. Αυτά λοιπόν είναι όλα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και ελπίζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μην προβάλλει ένσταση στην έγκριση της ε, κατεξότησης αυτής πράξης. Ευχαριστώ πολύ για τις διευκρινήσεις. Η κυρία, η κυρία Γκούτραντ ζητεί το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, ήρθα από άλλη συνεδρίαση και καθυστέρησα. Το θέμα όμως είναι πολύ σημαντικό και θέλω να μιλήσω γι' αυτό. Ιδιαίτερα επειδή γνωρίζω ότι στην ομάδα μου των σοσιαλιστών ανησυχούμε ε, για την πρόταση αυτή της Κομισιόν για ε, κατεξουσιοδότηση πράξη. Ε, υπάρχουν πολλές ανησυχίες σχετικά με τις επιπτώσεις στην υγεία. Πρέπει να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα ακριβώς. Εξετάζουμε μια ουσία η οποία υπήρχε, υπάρχει πολύ καιρό στο περιβάλλον αφού απορριφθεί, μπορεί να επηρεάσει τα οικοσυστήματα, διατηρείται, μπορεί να διδύσει στα ύδατα μέσα από τα φυτά και τα ψάρια, επανέρχεται στην τροφική μας αλυσίδα και ξέρουμε ότι στον άνθρωπο ε, πλήττει τα νεφρά, είναι πολύ επικίνδυνη ουσία που ε, μπορεί να είναι και καρκινογόνος και ξέρουμε και ότι η οστεοπόρωση επίσης μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά από το κάδμιο. Αφού τα ξέρουμε όλα αυτά και τα έχουμε κατανοήσει και επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να αντιπαλέψει με προηγούμενες εκπομπές γιατί πληττόμεθα από εκπομπές που ήδη πλέον υπάρχουν στο περιβάλλον πρέπει να ε, ε, ε, ε είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί να αντιμετωπίσουμε αυτό το τοξικό προϊόν για την υγεία και το περιβάλλον. Πρέπει να πω ότι στην πρόταση αυτή για την παράταση ε, πρέπει να πω ότι υπάρχουν διαθέσιμες νέες τεχνολογίες. Πιστεύω ότι η Κομισιόν δεν ε, τους δίνει τη δυνατότητα να εφαρμοστούν και αυτό είναι δυστύχημα. Και είναι και απογοητευτικό. Δεν εκπροσωπείται μαζικά η ομάδα μου εδώ, αλλά ξέρω ότι έγινε μια πολύ έντονη συζήτηση για αυτό το θέμα ακριβώς. Και η Κομισιόν προφανώς πρέπει να περιμένει ότι πολλές θα είναι οι δυνάμεις που θα αντιταχθούν σε αυτό που πάει να κάνει εδώ το λέω αυτό για να απαντήσω στην Κομισιόν. Θα γίνει σκληρή μάχη εδώ. Η Κομισιόν και μετά ο κύριος Τέιλορ αν θέλει να κλείσει τη συζήτηση αφού δοθήγουν διευκρινήσεις από την Κομισιόν. Ε, um, Ευχαριστώ πολύ για τα ενδιαφέροντα αυτά που είπαν οι συνάδελφοι. Να απαντήσω στην Κομισιόν. Είπατε ότι η γενική εξαίρεση ισχύει από 17 Ιουνίου μέχρι τον Ιούνιο του 17 κοντά στην ημερομηνία που θα εφαρμοζόταν αν είχατε ανακαλέσει την εξαίρεση τώρα επειδή υπάρχει περίοδος χάριτος πρέπει να δώσετε 12 με 18 μήνες. Αλήθεια είναι ότι τώρα έχουμε διαφορά μόνο 6 με 12 μήνες. Αλλά αυτό δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη χορήγηση μιας εξαίρεσης κατά των διατάξεων του νόμου. Άσε που μπορεί να είναι μεγαλύτερο το διάστημα από 6 με 12 μήνες αν δεχτείτε νέες εφαρμογές μέχρι το τέλος του χρόνου. Και ακόμα και αν αποφασίσετε να ανακαλέσετε την εξαίρεση, μπορεί να πάρει 18 μήνες μέχρι 18. Αν βάλετε και τα 12 με 18 μήνες περίοδος χάριτος, ε, είμαστε πια στο, στα μέσα ή στο τέλος του 2018. Αυτή η εξαίρεση προβλέπεται να λήξει τον Ιούνιο του 2018. Κα οποιαδήποτε εταιρεία που πιστεύει ότι έχει καλύτερη εναλλακτική μπορεί βεβαίως να υποβάλει μία πρόταση για την ανάκληση της εξαίρεσης ανα πάσα στιγμή. Συνάδελφοι, κοιτάζοντας ε, την αρχική πρόθεση της οδηγίας ΡΟΣ που ήταν να περιορίσει, να μειώσει τις βλαβερές ουσίες στον ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, νομίζω ότι αυτή η πρόθεση υπονομεύθηκε γιατί επετράπει ποσότητα καδμίου στο περιβάλλον μας ε, να αυξηθεί. Ε, στην ποσότητα του καδμίου να ε, αυξηθεί, γιατί αυτό σημαίνει η παράταση της ε, εξαίρεσης. Και τώρα μας κοιτούν οι ψηφοφόροι μας και οι πολίτες για να τους καθοδηγήσουμε. Η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δώσει ένα σίγουρο περιβάλλον για τους κατασκευαστές. Πρέπει να σας πω ότι εδώ έχω μια προσφορά ε, ε, ποσού 3.199 ευρώ που θα μπορεί να ε, παραδοθεί μέσα σε τρεις μέρες. Μπορώ να σας δώσω και έχει δηλαδή τεχνολογία καδμίου με κβαντικές κουκίδες. Υπάρχει τεχνολογία και μπορεί να την πάρετε και μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Ε, ε, εμείς πρέπει να, παρα... να, να τηρούμε την ε, κειμένη νομοθεσία. Τα κριτήρια για την επέκταση ή χορήγηση της παρέκκλησης σήμερα δεν πληρούνται και θεωρώ ότι η Κομισιόν πρέπει να επανεξετάσει την κατάσταση τώρα και όχι να προχωρήσει σε μια αδικαιολόγητη εξαίρεση. Πρέπει λοιπόν εμείς να απορρίψουμε την κατεξουσιοδότηση πράξη. Ε, θα προσθεθεί στην επόμενη Ολομέλεια μια πρόταση ψηφίσματος από την πλευρά μας και καλώ όλες τις πολιτικές ομάδες να την, να το, την προσυπογράψουν. Ευχαριστώ. Okay. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Οπότε εδώ ολοκληρώνω τη συνεδρίασή μας. Η επόμενη συνεδρίαση θα λάβει χώρα την 18η Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Στασβούργο και επόμενη στις 26 Μαΐου στις Βρυξέλλες. Ευχαριστώ πολύ και καλή σας όρεξη. Γεια σας.